So, we are going to start our committee meeting. Uh, welcome to... Ξεκινούμε λοιπόν τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλώς ήρθατε κυρία Κυριακίδου. Έχουμε τρία ζητήματα, ε, καυτά ζητήματα στη μέσα διάταξη σήμερα. Δεν θα, θα τα πούμε σειρά προτεραιότητας. Κορονοϊός, καρκίνος και ε, η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Ε, λοιπόν, πρώτα η Επίτροπος και μετά οι συγητές και μετά οι υπόλοιποι μιλητές. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις, ε, έχουμε ήδη 10 λεπτά καθυστέρηση, οπότε παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο που σας αναλογεί. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής ΕΝΒΗ, και Πρόεδρε, Σας βλέπω τόσο συχνά κάποιους από εσά που θα μπορούσα να σας αποκαλούμε το μικρό σας. Ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η καλή συνεργασία τα επόμενα πέντε χρόνια. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, και δεν το λέω ελαφρά την καρδία, η ανταλλαγή απόψεων, η συνή συνεργασία με το Κοινοβούλιο είναι εξαιρετικά σημαντική. Και αυτό γνωρίζω ότι είναι σημαντικό για όλους. Όλοι θέλουμε να πετύχουμε κάποια πράγματα ως Κοινοβούλιο, ως, Ευρωπαϊ... ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήμουν και βουλευτής για πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η συνεργασία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους μας τίμησαν με την παρουσία τους στην συνεδρίαση, στην, μάλλον στην στο δρόμενο της 4 Φεβρουαρίου όταν και παρουσιάσαμε το σχέδιο για τον καρκίνο ε, στείλαμε εκεί ένα πολύ ηχηρό μήνυμα ότι εμείς ως Ευρώπη θέλουμε να αναλάβουμε δράση κατά του καρκίνου. Μια δράση που να κάνει τη διαφορά. Και ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετείχαν, αλλά κυρίως η ενέργεια ε, που έβγαινε από τη συνάντηση αυτή, ε, έδειξε ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική βούληση αλλά και δημόσια υποστήριξη με τέτοια πρωτοβουλία. Ο άλλος τρίτος σημαντικός λόγος ε, για τον οποίο θεωρώ ότι αυτή η εκδήλωση ε, στέφθηκε από επιτυχία είναι ότι απέδειξε ότι παίρνουμε στα σοβαρά τους πολίτες, τους εμπλεκόμενους φορείς, τους επόμενους μήνες, όπως ξέρετε, ε, η στρατηγική αυτή είναι πολύ σημαντική για μένα και για πολλούς άλλους ε, σε αυτή την αίθουσα βέβαια, για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουμε φτάσει τώρα στην φάση του διαλόγου, της διαβούλευσης. Εσείς συμμετέχετε στη διαδικασία αυτή, θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να μοιραστείτε αυτές τις συζητήσεις με τους ε, ε, ψηφοφόρου σα με τι εκλογικέ περιφέρειε. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε όσο γίνεται περισσότερου ανθρώπου σε αυτή τη διαδικασία. Διότι αν δεν είναι συμπεριληπτική διαδικασία, αν οι άνθρωποι δεν νιώσουν ότι συμμετέχουν, δεν πρόκειται να σταθεί από επιτυχία το εγχείρημα. Κανεί δεν μπορεί να θεωρείται ιδιοκτήτη μια στρατηγική ε, κατά του καρκίνου. Είμαστε όλοι συνειδιοκτήτες ε, αυτής της στρατηγικής. Προσπαθούμε βεβαίως να εντοπίσουμε τις πιο σημαντικές δράσεις που πρέπει να λάβουμε εξετάζοντας ε, το όλο φάσμα από την έγκαιρη διάγνωση, την πρόληψη, ε, την περίθαλψη, τις γνώσεις, τον, τις νέες στον τομέα της έρευνας. Εξετάζουμε ε, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση λόγω των προβλημάτων που προκύπτουν με τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας. Βλέπουμε νέους ανθρώπους ε, οι οποίοι μπόρεσαν να επιβιώσουν από ένα ε, καρκίνο στην παιδική του ηλικία και που αντιμετωπίζουν διακρίσεις ε, λόγω αυτής της εμπειρίας τους στην επαγγελματική τους ζωή. Αυτό έχει να κάνει και με άλλες προτεραιότητες της Ένωσης. Υπάρχει και μια αποστολή έρευνας για τον καρκίνο στα πλαίσια του Οριζόντα Ευρώπη. Το Farm to Fork, όλα αυτά συνδέονται και με τη στρατηγική για τον καρκίνο. Πρόκειται για μια ενισχυμένη ενιαία πολιτική στον τομέα της υγείας. Θέλουμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, μια σφαιρική προσέγγιση και ειλικρινά νομίζω ότι εδώ μας δίνεται μια ευκαιρία ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εσείς έχετε κάνει πολλή δουλειά, έχετε, το έχετε αναδείξει ως προτεραιότητα, υπάρχει και η ομάδα των Ευρωβουλευτών κατά του καρκίνου, είναι πάνω από 100 άτομα σε αυτήν την ομάδα. Ε, εδώ και χρόνια λοιπόν έχετε αναδείξει το ζήτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον αποτελεί πολιτική προτεραιότητα και νομίζω ότι έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε το πρόσωπο του καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζω να το πετύχουμε. Ταυτόχρονα, το ανέφερε και ο Πασκάλ, εργαζόμαστε σκληρά ε, γύρω από τη στρατηγική ε, from Farm to Pork, από το αγρότημα στο πιάτο, ήταν και μέρος του Green Deal. Αυτό θέλαμε το Μάιο να το υποβάλουμε. Ε, τελικά το Μάρτιο όμως ε, θα το παρουσιάσουμε νομοθετικές και μη νομοθετικές προτάσεις θα περιλαμβάνει για να βελτιωθεί η βιωσιμότητα της διατροφικής αλυσίδας. Θα πρέπει να πάμε προς ένα διατροφικό σύστημα το οποίο θα είναι πιο ουδέτερο, πιο βιώσιμο, πιο θετικό σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτε θα έχουν ένα υψηλό επίπεδο διατροφική ασφάλεια. Αυτό δηλαδή που αναμένουν από εμά. Δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε όπω το παρελθόν και το εννοώ αυτό. Δεν το δέχονται οι πολίτε. Δεν δέχονται οι πολίτε το που συμβαίνει εδώ και αρκετά χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα περιβάλλον διατροφικό το οποίο είναι προσβάσιμο προς τους πολίτες να έχουν τις πληροφορίες στη διάθεσή τους και να μπορούν να τι καταλάβουν. Ε, πρέπει ταυτόχρονα να καταλάβουμε και να λάβουμε υπόψη μας τις ευρύτερες υπηρεσίες ε, των γεωργών, των αλλιέων που παράγουν τα τρόφιμα αυτά ε, που προφυλάσσουν τους ωκεανούς μας. Ε, πρέπει να φροντίσουμε να μην μείνει κανείς εκτός λοιπόν. Παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μετάβαση. Πρέπει να βρούμε τρόπο να τους υποστηρίξουμε. Η στρατηγική θα αφορά μια σειρά από προτεραιότητες μεταξύ των οποίων η μείωση της χρήσης των ε, ζενιοκτώνων, ε, ε, των χημικών, των αντιβιωτικών, των λιπασμάτων. Δεν θα μπω τώρα σε θα σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσει από αυτού. υπάρχουν σημαντικέ ανησυχίε των πολιτών και θέλουμε πραγματικά να, μπορέσουμε να προωθήσουμε ρεαλιστικού στόχου αλλά και δράσει. Θέλουμε να βελτιώσουμε την ενημέρωση του καταναλωτή σε ό,τι αφορά την επισήμανση των τροφίμων τα ζητήματα που προκύπτουν με τα απορρίμματα, τη σπατάλη δηλαδή τροφίμων και βεβαίως υπάρχει το θέμα από το αγρόκτημα ε, στο πιάτο, υπάρχει το θέμα της ευημερίας των ζώων, ένα θέμα που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Για να στηρίξουμε αυτή τη μετάβαση, η κοινή γεωργική πολιτική αλλά η κοινή ελευτική πολιτική θα είναι εξαιρετικά κρίσιμα εργαλεία. Θα συνεργαστούμε λοιπόν στενά για τη στρατηγική αυτή μαζί σα για να εξασφαλίσουμε ότι θα οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα και ωφέλη για του ανθρώπου την οικονομία και το περιβάλλον. Ε, η Επιτροπή ΕΜΒΙ εδώ παίζει ένα σημαντικό ρόλο για να βρεθεί ένα σωστό σημείο ισορροπία. Θα είμαι ανοιχτό, θα είμαι ανοιχτή μάλλον, θα σα ακούσω τι απόψει σα σήμερα, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όσο γίνεται περισσότερα ερωτήματα. Πάντα θα είμαι στη διάθεσή σας όμως ε, και στη συνέχεια ε, για να ακούσω αυτό που έχετε να μου πείτε. Και σύντομα να σας ενημερώσω και για το COVID-19, όπως ονομάζουμε πλέον το κορονοϊό, ε, ήταν μια από τις μεγάλες προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε έτσι πολύ νωρίς. Έχουμε καθημερινές εξελίξεις, ό,τι και να λέμε λοιπόν αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει. Το μήνυμά μου στην έκτακτη Σύνοδο Υπουργών Υγείας ε, την περασμένη εβδομάδα ήταν ότι πρέπει να έχουμε μια ενωμένη απάντηση απέναντι στο φαινόμενο, μια συντονισμένη αντίδραση, ε, διότι ο ιός αυτός δεν έχει σύνορα και ούτε εμείς πρέπει να βάλουμε σύνορα στην περίπτωση αυτή. Ε, παρακολουθούμε λοιπόν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα κράτη-μέλη υπήρξε μια πολύ καλή απάντηση, ανταπόκριση από τα κράτη-μέλη και ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να είναι πιο έτοιμα. Ψάχνουμε ε, χρηματοδότηση για τον λόγο αυτό. Θα ε, ε προωθήσουμε δημόσιες προμήθειες για ε, εξοπλισμό προστατευτικό του προσωπικού ε, συνεργαζόμαστε βεβαίως και με την ECDC και με τον ΠΟΗ. Ε, χρηματοδοτούμε την έρευνα για το εμβόλιο και υποστηρίζουμε βεβαίως και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εξωτερικό μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Βοηθούμε και την Κίνα ε, με την αποστολή έκτακτων, έκτακτου ιατροφαρμακευτικού υλικού. Είχαμε, ανταποκριθήκαμε άμεσα προς το αίτημα της Κίνας και, από, και 18 τόνοι ε, δόθηκαν από την Ιταλία ε, στην, ε, στον Ερυθρό Σταυρό στην Κίνα. Πρέπει πραγματικά να συνεργαστούμε όλοι και με την Κίνα για να μπορέσουμε να ε, δαμάσουμε αυτόν τον ιό. θα πρέπει να πάμε και πέρα από τις χώρες της Ένωσης, δηλαδή, στην προσπάθειά μας αυτή. Το COVID-19 είναι για μας ένα σαφές παράδειγμα της σημασίας της ε, σύμπραξης που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είμαι ικανοποιημένη ως Επίτροπος, διότι έως τώρα αυτό το επίπεδο συντονισμού, το συντονισμού ήταν καλό. Ε, επειδή όμως είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται καθημερινά, θα πρέπει όταν μιλάμε να έχουμε πάντα κατά νου ότι μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν εντός των επόμενων εβδομάδων. Αυτά δεν ξέρω αν ξεπέρασα τα 10-15 λεπτά που μου είχατε διαθέσει. Ευχαριστώ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε με το συντενιστή του ΕΛΚ, τον Πίτερ Λίζε. Στην οθόνη δεν φαίνεται, δεν αναγράφεται ο χρόνος. Θα σας καθοδηγώ λοιπόν εγώ όσον αφορά το χρόνο αγόρευσης. Θα σας ειδοποιώ όταν πλησιάζετε τα δύο λεπτά. Πρώτος λοιπόν ο Πίτερ Λίζ εξ του ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ καταρχήν για την εξαιρετική εκδήλωση πριν από δύο εβδομάδες στην αίθουσα της Ολομέλειας. Όπως είπατε κι εσεί βγήκε πολύ ενέργεια από αυτή τη συνάντηση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να την διοχετεύσουμε σε πραγματική δράση. Στο κέντρο των προσπαθειών μας πρέπει να είναι ο ασθενής, η ασθενής. Και στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να πετύχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τον καρκίνο και η επιβίωση να βελτιωθεί, να μπορέσουμε να καταγάγουμε νίκη κατά του καρκίνου δηλαδή. Οι ασθενείς ε, είπα πρέπει να είναι στο επίκεντρο αλλά και οι νομικοί πρέπει να μας συμβουλέψουν τι δυνατότητες έχουμε σύμφωνα με τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πού πρέπει να είμαστε λίγο πιο επιφυλακτικοί. Γιατί δεν θέλω στο τέλος να δώσουμε πολλές ε, συστάσεις στα κράτη-μέλη, χωρίς όμως να έχουμε μηχανισμούς για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει περισσότερα δεν, η Ευρώπη μπορεί να κάνει πράγματα ε, στο τομέα της υγείας. Με βάση τις, συνθήκες, τις, ε, ρυθμίσεις στην εσωτερική αγορά περιορίσαμε το γαπνό ε, πράγμα που μπόρεσε να γίνει. Δεν ήταν μόνο θέμα κρατών μελών λοιπόν. Και επίσης θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και για τους καρκινοπαθείς. Ε, έχουμε μια όξυνση της ε, κατάστασης σε ό,τι αφορά την έλλειψη των φαρμάκων. Αυτό προϋπήρχε ως κατάσταση, αλλά με τον κορονοϊό ε, επιδεινώνεται η κατάσταση. Θα ήθελα λοιπόν να πω στην Κομισιόν κατεπηγόντως να φροντίσει αυτό το θέμα κατά προτεραιότητα. Κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, φτάστε σχεδόν τα δύο λεπτά. Γιούτε. Πω πω μου ασκεί πίεση τώρα κατά αυτόν τον τρόπο, Πίτερ. Ευχαριστώ πάντω, Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για την παρουσίασή σας. Καταρχάς θα ήθελα να σα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ για τη δέσμευση και την προσήλωση που δείχνετε όσον αφορά την καταπολέμηση του καρκίνου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τη μάχη αυτή και πρέπει να σας πω ότι η δήλωση που κάνατε για τον κορονοϊό είναι ιδιαίτερη αξίας και θα ήθελα για μία ακόμη φορά να πω αυτό το οποίο λένε όλοι. Πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα, θα πρέπει να ανταλλάσσουμε μεταξύ ημών πληροφορίες. Τα όσα κάνετε είναι πάρα πολύ θετικά όσον αφορά την ε, πρόοδο, την εξέλιξη της επιστήμης. Χρειαζόμαστε τα επιστημονικά δεδομένα και την έρευνα. Και σε σχέση πάντως με τις τρίτες χώρες θα πρέπει να είναι σταθερή η θέση μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να ενημερωνόμαστε και να είναι έτοιμοι και οι Υπουργοί Υγείας μας. Τούτο λεχθέντον επιτρέψτε με να επιστρέψω στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, ένα σχέδιο ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, θα ήθελα να γνωρίζω πώ αντιμετωπίζετε τα αίτια του καρκίνου και σκέφτομαι για παράδειγμα εδώ πέρα τα ενοπνευματόδη ποτά, το αλκοόλ και τη διασύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον αυξημένο αριθμό των κρουσμάτων καρκίνου και την ε, καθημερινή έκθεση σε ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η DG Growth πρόκειται να συνεργαστεί με τη DG Envy για το ζήτημα αυτό, ιδίως όσον αφορά την επικείμενη ε, στρατηγική όσον αφορά τη μη χρησιμοποίηση χημικών ουσιών για τη βιωσιμότητα. Επίσης, όσον αφορά τις επιζήμιες ε, και οριζόντιες επιπτώσεις που έχουν οι χημικές ουσίες και κυρίως οι ονδοκρινικοί διαταράκτες. Μήπως θα έπρεπε εδώ πέρα να συνδυάσουμε τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς αντιμετωπίζει τελικά οριζόντια τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα πραγματικό ζήτημα υγειονομικό για την Ευρώπη αυτό. Όταν βλέπουμε ότι όλο και περισσότεροι πολίτες μας ζημιώνονται, ουσιαστικά βλάπτονται εξαιτία των ουσιών αυτών, εξαιτία των ενδοκρινικών διαταρακτών. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Εξ ονόματος της ομάδας Renew Europe θα μιλήσω γαλλικά, κυρία Επίτροπε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προαλήσαντες και να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που ξεκινήσατε τη δημόσια αυτή διαβούλευση όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στι 4 Φεβρουαρίου. Θέλετε πραγματικά πόσο κινητοποιημένοι είναι ορισμένοι ευρωβουλευτέ και ιδίω οι ευρωβουλευτέ που συμμετέχουν στην ομάδα κατά του καρκίνου, MEPS Against Cancer. Αναφερθήκατε στι πολύ μεγάλε προτεραιότητε, πρόληψη, ποιοτική φροντίδα και θεραπεία, έρευνα, ανταλλαγή δεδομένων, επανένταξη στο χώρο εργασία, παρηγορητική φροντίδα και ούτω καθεξής. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας θέσω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα σήμερα και θα ήθελα στο πλαίσιο αυτό της διαβούλευσης να σας μιλήσω για χρήματα. Το πρώτο μου ερώτημα έχει να κάνει με το βασικό αυτό άξονα της μάχης, τη χρηματοδότηση δηλαδή. Επί του παρόντος μπορείτε να μας πείτε ποιοι θα είναι οι βασικοί πόροι χρηματοδότησης όσον αφορά αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Στη δική μας Επιτροπή είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει τροπολογία στον κοινοτικό προπολογισμό σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό προκειμένου να βρεθεί κατάλληλη χρηματοδότηση. Τι έχει γίνει από αυτού. Στο πλαίσιο των ε, συζητήσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ποια είναι η άποψη που έχετε όσον αφορά την προβλεπόμενη χρηματοδότηση. Προβλέπετε κάποιο προκατακτικό εκτιμόμενος προπολογισμό για να χρηματοδοτηθεί αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Και μια δεύτερη ερώτηση. Πώς ε, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη κατανομή των προτεραιοτήτων όσον αφορά την αποστολή για την καταπολέμηση του καρκίνου από τον ορίζοντα Ευρώπη και ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Πρόκειται εδώ πέρα να έχουμε μια παράλληλη εξέλιξη και επεξεργασία των διαφορετικών προτάσεων. Ένα λεπτό και 53 δευτερόλεπτα. Λαμπρά, λέει ο πρόεδρο. Εξ ονόματος του ID Μάρκο Ντρεστό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρία Κυριακίδου επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της παρέμβασής σας ότι θέλετε να βοηθήσετε τους καταναλωτές να κάνουν τεκμηριωμένες συνειδητές επιλογές όσον αφορά τα υγιεινά τρόφιμα. Συμφωνούμε προφανώς με την πρόταση αυτή, αλλά πολύ φοβόμαστε ότι ο στόχος αυτός ενδεχομένως να μεταφραστεί τελικά σε συγκεκριμένε υποχρεώσει που θα επιβαρύνουν τους εθνικούς παραγωγούς και θα ε, ζημιώσουν τελικά τις εξαγωγές Ευρωπαϊκής Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε επισήμα των τροφίμων στο μπροστινό τμήμα των συσκευασιών που να δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες στου καταναλωτές. Αλλά αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί επισήμω. Επίση, έχουμε και το πρόγραμμα Nutri-Score το οποίο παρουσιάστηκε ως μοναδικό σύστημα εμπρόστιας επισήμασης των τροφίμων. Το σχέδιο αυτό δεν συνάδει όμως με το άρθρο 35 της, του αρμόδιου κανονισμού, του σχετικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθότι δεν δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά τη θρεπτική αξία των προϊόντων. Επίσης, δεν δίνει την πραγματική, τις πραγματικές ουσιαστικές πληροφορίες όσον αφορά τα τρόφιμα. Χρειαζόμαστε πραγματικά συνεκτικούς κανόνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση για να καταφέρουμε τελικά να προστατεύσουμε του καταναλωτέ εκείνου οι οποίοι θέλουν να έχουν συγκεκριμένε πληροφορίε. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να αποδεχθούμε ένα συγκεκριμένο σύστημα, το Nutri-Score, το οποίο μα επιβάλλεται εκ των άνω, ενώ υπάρχουν πολλοί άλλα συστήματα πέρα από το γαλλικό που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Το Nutri-Inform Battery, για παράδειγμα, το οποίο προτείνει η Ιταλία, όπου η θρεπτική αξία και οι υπόλοιπε πληροφορίε δεν παρουσιάζονται μόνο με χρώματα, ούτε υπάρχει μια αξιολόγηση θετική ή αρνητική, αλλά υπάρχει μια πιο ουδέτερη παρουσίαση των συστατικών, καθώς επίσης και των χαρακτηριστικών των τροφίμων και επιτρέπεται κατά αυτόν τον τρόπο στον καταναλωτή να πάρει μια αντικειμενική αμερόληπτη απόφαση. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν επιβάλλεται μονομερός μια άποψη όσον αφορά την θρεπτική αξία των τροφίμων. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να, έπρεπε, να έχει γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου προτού επιλεγεί το Nutri-Score. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιβληθεί ένα και μοναδικό μοντέλο όπω είναι το Nutri-Score το οποίο περιορίζει τελικά τις δυνατότητες των καταναλωτών να μερώνται σωστά. Για τους πρασίνους τώρα. Επίτροπε, ανα, μιλάτε ε, σχετικά με το Farm του Fork ότι η θερμοκρασία δεν μπορεί να μείνει σε αποδεκτά και ασφαλή επίπεδα εκτός και αν αλλάξει η παραγωγή τροφίμων. Χάρηκα που το είδα αυτό, αλλά δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να λέτε ότι η μελλοντική ΚΑΠ θα δώσει κίνητρα στους αγρότες να συμβάλλουν ενεργά στους κλιματικούς στόχους και ότι η στρατηγική Farm to Fork θα συμπληρώνει και θα στηρίζει απλώς τις προσπάθειες αυτές ε, συμμετέχω στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ Ευρωβουλευτής και φοβούμαι ότι πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι υπεραισιόδοξο και η διατύπωση έχει αλλάξει. Η νέα ΚΑΠ παραμένει business as usual σε μεγάλο βαθμό. Δεν έγινε αλλαγή μοντέλου ε, όπως ζήτησαν οι αγρότες και οι πολίτες. Και τέλος, η τελευταία έκθεση IPCC ε, λέει ότι χρειάζονται όλα αυτά. Και στην προηγούμενη κάπου υπήρχαν μέτρα για να ενθαρρυνθούν οι αγρότες να μειώσουν τις εκπομπές και να προστατέψουν το περιβάλλον. Οι εκπομπές το 2017 από τη Γεωργία ήταν στο ίδιο επίπεδο όπως το 2005 η βιοπικιλότητα, η ποιότητα του αέρα του εδάφους μειώθηκαν και οι μικροί, μικροί κλήροι, οι μικροί αγρότες μειώθηκαν ανησυχητικά. Η ΚΑΠ λοιπόν φαίνεται ότι δεν λειτουργεί ούτε για το περιβάλλον του ίδιου τους αγρότες. Το Farm to Fork δεν έχει νόημα αν παραμείνει μόνο στρατηγική χωρίς επιρροή στη, στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ. Ε, θα πρέπει επίσης να δούμε και την κοινή πολιτική αλληλείας ε, για τη βιοπικιλότητα χρειάζεται συστηματική αλλαγή. Το farm to fork, δευτερόλεπτα ζητάω, η farm to fork θα πρέπει να συνδυάζεται με την πράσινη συμφωνία και τους φιλόδοξους στόχους της. Και πώς γίνεται αυτό χωρίς σωστή οικολογική αξιολόγηση της ΚΑΠ. Η ενωσιακή πολιτική αυτή ε, ε, ε, παίρνει το μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Και πόσο μακριά είστε διατεθειμένοι να πάτε στις αναλύσεις σας του συστήματος τροφίμων. Θα πιέσετε ώστε να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές. Συγγνώμη που μακρηγόρησα, ευχαριστώ. Για το ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. τον χάρτη πορείας για την καταπολέμηση του καρκίνου, τον μελέτησα πολύ και συμμετείχα και στην εκδήλωση που αναφέρατε στην αρχή. Η... Τρόποι καταπολέμησης του καρκίνου, δηλαδή διάγνωση, πρόληψη, ε, θεραπεία, ε, μετέπειτα θεραπεία, παρηγορητική κλπ. Ε, όλα αυτά συνάδουν και με την πολιτική που ακολουθούμε στην Πολωνία. Ε, πρόσφατα ε, εγκρίναμε το σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου και της αντιμετώπισης των ασθενών όπου ο ασθενής βέβαια βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο όλων αυτών των δραστηριοτήτων, των δράσεων. Η πρόσβαση στη θεραπεία πρέπει να είναι εξασφαλισμένη για όλους τους ασθενείς ανεξάρτητα από τον τόπο διαβίωσής τους. Τώρα, κάποιες ερωτήσεις που αφορούν κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το κέντρο ε, για τον καρκίνο. Πρόκειται εδώ για μεθόδους ερευνητικές, ε, έρευνες. Η ιδέα δημιουργίας μιας τέτοιας πλατφόρμας για τον καρκίνο μου φαίνεται πολύ καλή και υποστηρικτική της υλοποίησης των εθνικών στρατηγικών. Ρωτώ όμως, πόσο συγκεκριμένα έχουν διαμορφωθεί οι δραστηριότητες αυτού του κέντρου. Για παράδειγμα, η δομή έρευνας ε, σε όχι τόσο ε, πλούσια κράτη ε, ίσως δεν έχει ακόμα επαρκώς προετοιμαστεί όπως για παράδειγμα τον τρίτο πυλώνα του προγράμματος. Ίσως θα πρέπει επίσης να υπάρχει μια ίσαιο κατανομή των πόρων από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά την ιατροφαρμακευτική υποδομή και άλλα θέματα. Και ερωτώ, κονδύλια και υποδομή για την καταπολέμηση του καρκίνου θα δοθούν σε ε, στο ίδιο επίπεδο και θα αλλάξουν μόνο οι επενδύσεις και οι ροές των επενδύσεων και επίσης ε, με τον ίδιο τρόπο οι δραστηριότητες, οι επενδυτικές θα συνεχιστούν. Και τέλος, Ποιες είναι οι προκλήσεις που δεν είναι οικονομικής φύσεως, αλλά όμως είναι προτεραιότητες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Για την ΚΟΕ, ο τελευταίος συμμιλητής σε αυτό τον γύρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι πολύ επίκαιρα τα θέματά σας. Αυτό το Σάββατο είναι η ε, ημέρα των σπανίων νόσων και διοργανώνονται διάφορες ε, δραστηριότητες ε, αυτή τη βδομάδα. Αναφέρατε την καταπολέμηση του καρκίνου. Υπάρχει όμως μεγάλο δυναμικό και για την έρευνα των σπανίων νόσων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει εδώ να αναδειχθεί σε ένα σύμβολο συνεργασίας, να καταφέρει να επιτύχει κάτι από κοινού. Θα μπορούσαμε να έχουμε ε, ε, εξυγχρονισμό νομοθεσίας. Μιλάμε για τη βοήθεια των ασθενών, ε, αλλά μπορούμε να τους βοηθήσουμε χάρη στην γρήγορη πρόσβαση στην υγεία και στη φροντίδα. Ε, αυτά θα πρέπει να εγκριθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου οι ασθενείς που έχουν είτε καρκίνο είτε κάποιο άλλο σπάνιο νόσημα να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουν όλοι αυτοί πρόσβαση στην υγεία. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούμε να προσφέρουμε θεραπεία παντού στην Ευρώπη. Καμιά φορά ασθενεί στη Γαλλία ή στη Γερμανία έχουν καλύτερη φροντίδα από ότι οι ε, ασθενείς στην Ανατολική Ευρώπη. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό και πώς θα προχωρήσετε στην θέσπιση νομοθεσίας που θα μπορέσει να βοηθήσει ε, να γίνει αυτό. Ε, Επίση ε, φαντάζομαι ότι και άλλοι συναδελφοί σας θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Υπάρχει ένα πακέτο για τον καρκίνο, η άλλη είναι το Farm to Fork, από το αγρόκτημα στο πιάτο δηλαδή. Και μετά θα συνεχίσω με τον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρώτο γύρο. Δεν ε, είμαι βέβαιη ότι μπορώ να τα βάλω σε δέσμες, γιατί την υγεία δεν την προσεγγίζω έτσι. Ούτε μπορούμε να τη δούμε έτσι. Το, δεν μπορεί να είναι ένα πακέτο το καρκίνος και ένα άλλο πακέτο να είναι το farm to fork, γιατί αν το δείτε έτσι γυρίζομαι σε προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν για πολύ καιρό. Uh, λοιπόν, θα αναφερθώ σε κάποια θέματα. Ίσως δεν απαντήσω σε όλα, αλλά μπορώ να επανέλθω. Καταρχήν, μια γενική αρχή. Από εκεί θα αρχίσουμε. Κάποιος είπε πολύ σωστά ότι πρέπει οι πολίτες και οι ασθενείς να είναι στο επίκεντρο της στρατηγικής μας. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και για σας όλους και για μένα ως Επίτροπο για την Υγεία και την Ασφάλεια Τροφίμων. Είναι προτεραιότητα. Έτσι πρέπει να δουλέψουμε. Αν δεν αρχίσουμε με καλή θέληση και αν δεν δεχτούμε ότι οι ασθενείς και οι πολίτες θα είναι στο επίκεντρο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τόσο απλά. Δεύτερο, τι θα κάνουμε, αν θα επικεντρώνουμε στους ασθενείς. Ε, αν μπορώ να κατηγορηθώ για κάτι, είναι ότι υπερβολικά βάζω τους ασθενείς στο επίκεντρο. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία όμως σε σχέση με το τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Ο Πέτερ Λίζε μίλησε για την ενέργεια που ήταν στην ε, έστουσα κατά την πρώτη μας εκδήλωση και ότι πρέπει να διοχετευτεί σωστά. Η αίσθηση που είχα μετά την εκδήλωση αυτή είναι ότι ναι, ήταν για πάρα πολύ ενέργεια και αυτό ήταν θετικό. Την επόμενη μέρα ξύπνησα με μια τρομερή αίσθηση της τεράστιας ευθύνης που έχουμε όλοι, γιατί οι προσδοκίες ανέβηκαν πολύ ψηλά σχετικά με τον καρκίνο και πρέπει εμείς να ανταποκριθούμε. Από την πρώτη μέρα λοιπόν αρχίσαμε. Ήδη έχουμε αρχίσει όχι μόνο να συναντώμεθα με τους εμπλεκομένους, αλλά και προσωπικά θα ενημερώνουμε κάθε δύο εβδομάδες και έχουμε κάθε μήνα συνάντηση για την πορεία του προγράμματος, για να βεβαιωθούμε ότι θα συνεργαστούμε όλοι για να γίνει το πρόγραμμα. Τώρα, η νομική ειδική και νομοθεσία, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το απαντήσω. Τα κράτη-μέλη έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά που συνεχίζεται και πρέπει να δούμε πού βρίσκονται τα προβλήματα. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε ενημέρωση από εσά. ευχαριστώ για τα σχόλια για τον κορονοϊό και το επίπεδο ετοιμότητας. Έχετε πολύ δίκιο. Γι' αυτό από την αρχή είπα ότι πρέπει να είμαστε προορατικοί. Κάθε φορά που έχουμε την ε, ε, κακή είδηση ενός κρούσματος στην Ευρώπη, ενημερώνω τον Υπουργό πριν φτάσει στο Συμβούλιο Υπουργών Υγείας. Ρωτώ τι έγινε, τι χρειάζονται. Αυτό σημαίνει προορατικός. Δεν πρέπει εκ των υστέρων να τρέχουμε και να λέμε θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει καλύτερα. Ε, βέβαια υπάρχουν σφάλματα σε αυτά που κάνουμε, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις όπως έρχονται. Υπό αυτή την έννοια πήγα, απευθύνθηκα σε κάθε Υπουργό Υγείας όταν είχαν επιβεβαιωμένα κρούσματα πριν από το Συμβούλιο Υγείας. Τώρα για το Farm to Fork το σχέδιο καταπολέμησης του καρκίνου και το ζήτημα των ενδοκρινικών διαταρακτών. Είπα στην αρχή ότι το σχέδιο κατά του καρκίνου και το Farm to Fork δεν θα διαχωριστούν. Πολλά από αυτά που είναι στο Farm to Fork θα πάνε στο σχέδιο για τον καρκίνο και αντίστροφα, γιατί πρέπει να δούμε θέματα που αφορούν την πρόληψη. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι ένα τεράστιο θέμα όπως γνωρίζετε. Πολλοί από εσά ε, στην αίθουσα αυτή έχουν περισσότερη πείρα από ό,τι εγώ. Αλλά όσο πιο πολύ διαβάζω, τόσο πιο πολύ μαθαίνω και τόσο πιο πολλά πιστεύω ότι χρειάζεται να ξέρω. Υπάρχει και ένα fitness check που γίνεται και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Έχουμε ήδη νομοθετήσει για τα ε, βιοκτώνα και τα ζυζανιοκτώνα, σημαντικό αυτό. Δεν είναι εύκολο να αξιολογήσουμε τους κινδύνους και η ΕΦΣΑ τώρα ε, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων δουλεύει εκεί. Θέλουμε να μπορούμε να αξιολογούμε τι γίνεται και με άλλα υλικά, με άλλες ουσίες, γιατί πολλές ανησυχίες αφορούν άλλες γενικές διευθύνσεις και όχι ε, που αφορούν παιχνίδια, ε, καλλιντικά κλπ. Και θα ε, υποβάλλουμε μια πρόταση για το Farm to Fork σε αυτά τα πλαίσια και επίσης προσπαθούμε να δούμε, και αυτό δεν είναι εύκολο, τους κινδύνους εις ό,τι αφορά τα λεγόμενα cocktail effects. Όλα αυτά τα εξετάζουμε. Αρκετοί είπαν για τον καρκίνο σε σχέση με τη χρηματοδότηση των μέτρων, η Βερονίκ. Έχετε δίκιο που ανησυχείτε γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν προγράμματα και όχι χρηματοδότηση. Αλλά αυτό είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν, οπότε υπάρχουν κονδύλια. Το είπε και η πρόεδρος Φοντερ Λάιν. Οπότε θα υπάρχει χρηματοδότηση μέσα από το Cancer Mission από το Horizon και την Cancer Mission η οποία θα εργαστεί με το Cancer Plan. Δεν θα δουλέψουμε χωριστά. Εκεί χρειάζεται το, η, η, η συμβουλή τους, η ενημερωσία τους. Υπάρχουν και από το Κοινωνικό Ταμείο και από τα ψηφιακά ταμεία γιατί η ηλεκτρονική, η ηλεκτρονική υγεία είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορώ να σας πω τώρα ακριβώς ποια θα είναι τα ποσά που θα δοθούν, αλλά μπορώ να σας πω ότι επειδή είναι προτεραιότητα της Κομισιόν αυτό το πράγμα, θα υπάρξει χρηματοδότηση επαρκή για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να εφαρμοστεί η στρατηγική κατά του καρκίνου. Υπήρχε μία ερώτηση ε, και από μια, μια ε, Ιταλίδα συνάδελφο για, το, για τη σήμανση. Το Farm to Fork θα μιλήσει και για το, ε, τη σήμανση, επισήμανση, αλλά πρέπει να δούμε τη βασική αρχή εδώ. Όλοι πρέπει να το δούμε αυτό. Η βασική αρχή είναι ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να παίρνουν ξεκάθαρες πληροφορίες για το τι αγοράζουν από το ράφι. Δεν θα μπορέσω να σας πω τώρα ποια θα ε, είναι αυτή η ενημέρωση. Τώρα θέλουμε να δούμε ε, τη βαθμολογία, ε, κάποιο σύστημα σήμανσης. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τις διαδικασίες, γιατί έτσι θα έχουμε καλύτερες πληροφορίες. Υπάρχουν ανησυχίες σε κάποια κράτη-μέλη σχετικά με το, την επισήμανση και πώς θα είναι. Όλα θα αξιολογηθούν και στα πλαίσια του προγράμματος Farm to Fork θα υποβάλουμε μια πρόταση. Οπότε ε, το αφήνω το θέμα προς το παρόν εδώ. Για την ΚΑΠ, Πράσινη Συμφωνία και ΚΑΠ. Δίκιο έχετε. Υπάρχει ανησυχία σχετικά. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Η ΚΑΠ πρέπει να είναι φιλόδοξη και να καλύπτει και να εφαρμόζει τις προτάσεις της Πράσινης Συμφωνίας, Green Deal. Τώρα κάνουμε μια ανάλυση που ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πώς η ΚΑΠ μπορεί να ανταποκριθεί στις ε, φιλοδοξίες του Green Deal, της Πράσινης Συμφωνίας. Θα επανέλθουμε. Κάποιος ρώτησε αν θα πιέσω. Θα, ε, ναι, θα πιέσω. Εγώ είμαι επίτροπο για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων. Αυτό είναι ο τίτλος, αλλά είναι και η προσωπική μου πεποίθηση, το ήθο μου. Ναι, προχωράμε, το Farm to Fork θα είναι φιλόδοξη στρατηγική, θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά εγώ βρίσκομαι εδώ για να προστατεύσω τους καταναλωτές και θέλω να ανταποκριθώ σε όσα αναμένουν από μένα. Τώρα για τις σπάνιες νόσους. Υπάρχει μια εκδήλωση του Κοινοβούλιο εδώ δεν θα μακρηγορήσω πολύ ακόμα. Ε, να ένα παράδειγμα τι μπορούν να κάνουν οι ευρωβουλευτέ μαζί. Ε, εδώ υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς. Αυτά, υπάρχουν δίκτυα αναφοράς. Και εκεί, από εκεί μπορούν οι ασθενείς να ε, ενημερωθούν. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ε, υποστηρίξουμε. Είναι ένα σύμβολο του τι μπορούμε να πετύχουμε μέσα από τη συνεργασία και πολλά περισσότερα μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, μιλήσατε για την ε, αξιολόγηση της ε, τεχνολογίας για την υγεία. Ε, υπάρχουν προβλήματα εδώ, δεν προχωράει πολύ καλά, δεν το υποστηρίζουν όλα τα κράτη-μέλη και όλοι οι εμπλεκόμενοι. Εδώ μπορείτε εσείς ως ευρωβουλευτές να βοηθήσετε μέσω του των κρατών μελών σας για να εξασφαλιστεί η υποστήριξη. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε με την πρόταση αυτή της Κομισιόν. Αυτή η αξιολόγηση της τεχνολογίας υγείας είναι σημαντική για του ασθενείς. Πρέπει να προχωρήσει. Πώς θα γίνει αυτό, Εγώ άρχισα να θέτω το ζήτημα σε όλες τις διμερείς επαφέ με τους υπουργού, ιδιαίτερα ε, εκείνους που ξέρω ότι έχουν προβλήματα, όταν προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι το οποίο το είχαμε για πολύ καιρό, θα πρέπει να δούμε πού βρίσκονται οι ανησυχίες, οι επιφυλάξεις, να δούμε πόσο ευέλικτοι μπορούμε να είμαστε και η Κομισιόν ήταν ευέλικτη και πώς μπορούμε να διασκεδάσουμε τους φόβους τους για να προχωρήσουμε παραπέρα. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να το προχωρήσω. Επίσης περιμένουμε την αξιολόγηση ε, της ε, Νομοθεσία για τα παιδιατρικά θέματα που θα μας δώσει ε, απαντήσεις σε σχέση με κάποια φαρμακευτικά προϊόντα που είναι και αυτά κομμάτι της στρατηγικής μας. Λοιπόν, νομίζω ότι αναφέρθηκα στα περισσότερα. Όσο όσα δεν αναφέρθηκα μπορείτε να επανέλθετε. Ευχαριστώ. Ναι και βεβαίω έχετε δίκιο. Όλα τα θέματα συνδέονται μεταξύ τους παρότι δεν είναι πακέτο. Θα περάσουμε τώρα στο δεύτερο γύρο Έχετε ένα λεπτό ο καθένας πλέον. Θα είμαι αυστηρός, διότι είναι πολλά τα ερωτήματα. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε... Αν δεν μπορούμε να σας δώσουμε το λόγο, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίει η γραμματεία, αυτά είναι οι συντονιστές σας. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για σας πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ξεκινάμε από το ΕΛΚ, η Τζέσικα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Θα μιλήσω σου ειδικά. Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική από το αγρόκτημα ε, στο πιάτο, όλο το θέμα εδώ είναι η βιωσιμότητα. Και όταν μιλάμε για βιωσιμότητα, υπάρχει το θέμα της υπερβολικής χρήσης αντιβιωτικών στην Ευρωπαϊκή Γεωργία η εμπειρία από το παρελθόν μας δείχνει ότι αν θέλουμε μια νομοθεσία για, το, για ένα τέτοιο ζήτημα θα, θα πάρει πολύ χρόνο. Στη στρατηγική λοιπόν αυτή η Κομισιόν ποια μετάσκοπεύει να πάρει σε ό,τι αφορά τη χρήση αντιβιωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να είναι πιο βιώσιμη και η πρόσφατη νομοθεσία ε, για τα, για τα προϊόντα έχει πετύχει η Κομισιόν σκοπεύει να την καταστήσει πιο αυστηρή ή να νομοθετήσει εκ νέου εάν χρειαστεί. Παρακαλώ η Μυρία Μντάλη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Πίτροπε, ευχαριστώ και δημοσίω για την προσβασιμότητά σας και τον ανοιχτό σας, τον ανοιχτό σας πνεύμα. Τα ερώτημα πρώτα απ' όλα ε, για την καταπολέμηση του καρκίνου. Είπαμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα κοινό ε, χώρο δεδομένων ε, για την υγεία. Πώς θα λειτουργήσει αυτό, διότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν έχουν καν ένα εθνικό χώρο με δεδομένα για την υγεία. Συχνά υπάρχουν τα στοιχεία, αυτά τα δεδομένα αποθηκευμένα σε πλατφόρμες διαφορετικές και μη ε, συμβατέ μεταξύ του. Πώ μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι σκοπεύετε να κάνετε. Και επανέρχομαι σε ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα. Πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά να, να, ε, να φροντίσει έτσι ώστε τα σπάνια φάρμακα να είναι διαθέσιμα σε όλα τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση των σπάνιων ασθενειών εννοώ, ε, αλλά και τον καρκίνο. Πώ μπορούν να έχουν ε, δηλαδή εύκολη πρόσβαση στα χρώματα του οι Ευρωπαίοι όπου και να βρίσκονται. Ε, ευχαριστώ από τη Renew τώρα. Ευχαριστώ κύριε, κυρία Πέτρο που είστε εδώ σήμερα. Για τον COVID-19 ε, είναι αρκετά εντυπωσιακή αριθμή. Εγώ ως γιατρός πρέπει να σας πω ότι πάντα σκέφτομαι τους ανθρώπους με πίσω από τα νούμερα αυτά. Είναι εντυπωσιακό, αυτό που κάνουν οι Κινέζοι. Έχουν φτιάξει νοσοκομεία ολόκληρα μέσα σε λίγες μέρες και παρότι δεν γνωρίζουμε αν οι κινέζικες αρχές τα κάναν όλα σωστά, πρέπει να αναρωτηθούμε ε, πώς η Ευρώπη θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση. Βεβαίω και είναι σωστό ε, ένα μεγάλο μέρο των ζητημάτων υγεία να είναι εθνικό ζήτημα. Όμω χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη για κάποια ζητήματα όπω ε, η αδειοδότηση. Η ECDC χρειάζεται περισσότερε αρμοδιότητε και περισσότερου πόρου σε σχέση με τι ΗΠΑ. Ε, είναι πολύ φτωχ, φτωχή η ECDC. Επίσης, σε μια κατάσταση κρίσης ε, θα πρέπει η αχρίαστη γραφειοκρατία να μην ε, επιβραδύνει τις διαδικασίες. Θα πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνη η SEDC όχι μόνο για τις μελέτες σε φάσεις 3 αλλά και για τις φάσεις 1 και 2. Ιδιαίτερα όταν χρειαζόμαστε επιγόντως κάποια φάρμακα. Ποια είναι η θέση σας για αυτά τα δύο ζητήματα, ποια βήματα σκοπεύετε να πάρετε. Ε, λειτουργεί καλά η Ευρώπη στον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά μπορούμε σίγουρα να βελτιωθούμε. Για το ΕΛΚ και πάλι, κυρία Μονσεράτ. Ναι, ευχαριστώ πολύ, ε, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Σας συγχαίρω για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του, του καρκίνου και για την διαδικασία διαβούλευση, Ίσως ώστε οι εμπλεκόμενοι φορεί, οι ασθενεί, οι θεσμοί να συμμετάσχουν ε, με ένα συμπεριληπτικό τρόπο για να καθορίσουμε από κοινού τι προτεραιότητε. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στο θέμα τη πρόληψη. Ε, στην πρόταση του δικού χάρτη η πρόληψη θεωρείται ένας πολύ σημαντικός πυλώνας. Όταν όμως μιλάμε για πρόληψη, ορισμένες φορές ε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε την ψυχική υγεία. Το άγχος ε, δημιουργεί πολλές ασθένειες και μεταξύ των οποίων και τον καρκίνο. Θα πρέπει να, μάθουμε να διαχειριζόμαστε το άγχος, το στρες, καθώς και το ψυχολογικό άχθος που είναι ε, ε, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το επίπεδο κινδύνου και ρίσκου. Προσπαθούμε να προωθήσουμε ε, μια υγιή ζωή, μια υγιή τρόπο ζωής, υγιή διατροφή, καταπολέμηση του καπνίσματος. Πρέπει όμως να πάρουμε και μέτρα προλεπτικά και για την ψυχική υγεία. Το ευρωπαϊκό σχέδιο λοιπόν θα συμπεριλάβει μέτρα σφαιρικά ε, για την πρόληψη ε, της ψυχικής ιδέας ό,τι αφορά τον κίνδυνο καρκίνου. Madame le commissaire, monsieur le président. Κυρία Επίτροπε, ε, η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο καλύπτει το σύνολο της διατροφική αλυσίδα εξορισμού. Η, η, σχέση μεταξύ βιομηχάνων όμω και γεωργών ε, βρίσκει τους γεωργούς να μένουν απ' έξω στο τέλος. Ε, η μελτίωση των ελέγχων σε ό,τι αφορά το, το υγειονομικό κομμάτι τη διατροφική δεν πρέπει να δημιουργήσει κίνδυνο για τι μικρέ εκμεταλλεύσει και τι μικρέ βιομηχανίε. Γνωρίζουμε ότι συχνά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τι διαδικασίε συμβατότητα. Έχω λοιπόν δύο ερωτήματα να θέσω. Πώ μπορείτε να εγγυηθείτε ότι αυτή η στρατηγική δεν θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα 10 εκατομμύρια εκμεταλλεύσει μικρέ εκμεταλλεύσει στην Ευρώπη. Επίσης, πω μπορείτε να, να, να εγγυηθείτε ότι αυτή η στρατηγική δεν θα δημιουργήσει μειονέκτημα στις μικρέ στις ό,τι αφορά την συμβατότητα και δεν θα ενισχύσει τα βιομηχανικά μονοπόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την S&D τώρα ο κύριος... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, όπως αναφέρατε, οι πολίτες Θέλουν να ξέρουν τι αγοράζουν, τι τρόφιμα τρώνε. Δεν αφορά αυτό μόνο την ε, θρεπτική αξία, αλλά και την προέλευση. Και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς ενδεχομένους. Όλα αυτά δεν έχουν διευκρινιστεί επαρκώς. Το Κοινοβούλιο για τη Σόγια και την προέλευσή της έχει θέση. Απέρριψε την πρόταση δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα. Ε, οπότε η Κομισιόν πώς θα αντιμετωπίσει τις ε, ε, προτιμήσεις και θέσεις του Κοινοβουλίου. Θα σέβεται τις πλειοψηφικές αποφάσεις του Κοινοβουλίου και θα μπορέσει να προχωρήσει στην ε, ε, ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται. For, ε, για τους πράσινους. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ στην Επιτροπή μας Σα ευχαριστούμε για το πολύ φιλόδοξο αυτό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου που ξεκίνησε στι αρχέ του μήνα. Όσον αφορά την πρόληψη τώρα και πώ συνδέεται αυτή με τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Το συζητήσαμε αυτό και μα υποσχεθήκατε ότι ε, θα εργαστείτε προκειμένου να μειωθεί η χρήση των φυτοφαρμάκων κατά 50% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό είναι πολύ φιλόδοξο. Αλλά διαβάσαμε χθε σε πολλές εφημερίδες από το, το ότι υπάρχει μια έντονη πίεση από διάφορες επιχειρήσεις όσον αφορά τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων, τα οποία έρχονται αυτή τη στιγμή από εισαγωγές, από προϊόντα δηλαδή τρίτων χωρών. Πώς μπορείτε εσείς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιταχθείτε στις δυνάμεις εκείνες που θέλουν εμπορικέ συμφωνίες με μεγάλες επιχειρήσεις από τον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες ε, ουσιαστικά διατηρούν και ενισχύουν πολύ συχνά τις μεγάλες αυτές επιχειρήσεις στον τομέα των φυτοφαρμάκων. Σας ευχαριστούμε. Ας ακούσουμε τώρα και τις απαντήσεις. Συγκεκριμένες ερωτήσεις περιμένουμε και συγκεκριμένες απαντήσεις. Θα απαντήσω όσο καλύτερα μπορώ. Τώρα θα το κρίνετε εσείς αν είναι αρκετά συγκεκριμένες ή όχι. Πάντως θα είμαι εδώ πέρα μαζί σας και τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θίξατε, καταρχά γενικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Ω προ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται ένα νομικό πλαίσιο το οποίο έχει θεσπίσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αποφάσει αδειοδότηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για, τα, για, του τους έχουν να κάνουν με τι συστάσει τη ΕΦΣΑ. Και θα πρέπει κάθε φορά να πληρούνται βέβαια ε, οι διατάξει τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού. Θεωρώ ότι το σύστημα αυτό μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό. Είμαι διαλλακτική και ανοιχτή απέναντι στι δικέ σα τι προτάσει. Πάντω, μέχρι να γίνει αυτό, μέχρι να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προφανώ θα ακολουθεί του κανόνε προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ξέρετε ότι ήδη από το 2017 είχαμε πει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να επιλέξουν opt-out για άλλους λόγους πέραν της ασφαλείας, αλλά αυτό δεν εγκρίθηκε από τους συνομοθέτες δυστυχώς. Για τα αντιβιωτικά τώρα, τεράστιο το ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στο πλαίσιο του νέου αυτού προγράμματο για την υγεία οριζόντια. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε δηλαδή το ζήτημα των αντιβιωτικών, η χρήση αντιβιωτικών, η κατάχρηση μάλλον θα έλεγα αντιβιωτικών και το όλο ζήτημα της μικροβιακής αντοχής είναι τεράστιο ζήτημα. Προσπαθούμε να θεσπίσουμε κάποιους δείκτες τώρα για να μειωθεί το φαινόμενο αυτό. Υπάρχει επίσης ε, μια νέα νομοθεσία, μια νέα πρόταση νομοθεσίας που θα ισχύει από το 2022 και μετά όσον αφορά τα κτηνιατρικά φάρμακα και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί θα προσπαθήσει να ρυθμίσει τη χρήση αντιβιωτικών ε, στα ζώα αλλά βέβαια θα πρέπει να προσεγγίσουμε το ζήτημα αυτό και στα πλαίσια της φαρμακευτικής στρατηγικής. Οριζόντια λοιπόν θα πρέπει να αντιμετώπιση για το ζήτημα των αντιβιωτικών. Τώρα, όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων, Υγειονομικών Δεδομένων, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε εδώ ότι θα πρέπει να σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τα δεδομένα και την ψηφιοποίηση των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναφέρομαι στα υγειονομικά δεδομένα. Υπάρχουν κάποιε προκλήσει σε σχέση με τα δεδομένα υγεία. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί να υπάρχουν κώδικε διοντολογία, να υπάρχει μια συγκεκριμένη διακυβέρνηση Υπάρχουν ε, διάφορα σχέδια τα οποία μελετούμε αυτή τη στιγμή για να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε διαλειτουργικότητα μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί είπατε και εσεί ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία έχουν προχωρήσει περισσότερο από ό,τι άλλα. Ελπίζω πάντω ότι μέχρι το, τα τέλη του έτου θα είμαστε σε θέση να υποβάλουμε επίσημη πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, όσον αφορά το COVID-19. Ακούστηκαν και άλλε παρατηρήσει για τον κορονοϊό όσον αφορά την ε, συνεργασία, όσον αφορά την έρευνα. Θα ήθελα να σας πω ότι αμέσως μετά την έξαρση των κρουσμάτων αυτών αγκρίναμε νομίζω 10 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα πρέπει να δοθούν για την έρευνα που θα πρέπει να γίνει ειδικά για τον κορονοϊό για να αναπτυχθεί ένα νέο εμβόλιο. Και μάλιστα θα υποστηρίξουμε σαφώς την έρευνα στον τομέα αυτό. Είμαστε δεσμευμένοι ως προς αυτό. Η ψυχική υγεία Αν μιλάμε για υγεία ανθρώπινη, υγεία των ζώων και υγεία των φυτών, θα έλεγα ότι η ψυχική υγεία αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης υγείας. Δεν μπορούμε να δούμε κατακαιρματισμένα και απομονωμένα την σωματική υγεία από τη μία πλευρά και την ψυχική υγεία από την άλλη, αλλά μόνο από κοινού μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους δύο αυτούς τομείς και σαφώς η ψυχική υγεία μπορεί να επηρεάσει εν γέννη την ε, ανθρώπινη υγεία και αυτό το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολύ έντονα. Όσον αφορά τώρα τους ε, κανόνες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όταν ασκείται πίεση αυτή τη στιγμή από μεγάλες βιομηχανίες, διαβάζω και εγώ διάφορα άρθρα στον τύπο, αλλά προτιμώ να μην αναλώνομαι στην ανάλυση διαφόρων σενάριων. Οι εμπορικές πάνω συμφωνίες δεν αλλάζουν το επίπεδο ασφάλειας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ότι συναντιόμαστε με εκπροσώπους επιχειρήσεων δεν σημαίνει ότι πρόκειται να μειώσουμε τα πρότιμά μας όσον αφορά τον τομέα της υγείας και εγώ θα συνεχίσω να καταβάλω άοκνες προσπάθειες για να προστατεύσω την υγεία των καταναλωτών και το περιβάλλον τώρα. Το πώς θα το πετύχουμε αυτό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το να διαπληκτιζόμαστε, με το να βρισκόμαστε συνεχή αντιπαράθεση. Υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα στα οποία θα πρέπει να βασιστούμε και αυτά θα πρέπει ουσιαστικά να διέπουν και τα επιχειρήματά μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και θα είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη και όσον αφορά τη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο. Είναι πρωτόγνωρο το επίπεδο φιλοδοξία το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τι προτεραιότητε που θέτουμε για την υγεία των καταναλωτών και των περιβάλλων δεν πρόκειται να επαναχωρήσουμε στις βασικές μας αυτές προτεραιότητες. Και αν μου επιτρέπετε ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Πρόεδρε που μπορεί να μην είναι πάρα πολύ χειροπιαστό και συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να εργαστούμε οριζοντίως, διατομεακά. Και γι' αυτό το λόγο και η Επίτροπη, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, δεν θέλουμε να εργαζόμαστε πλέον απομονωμένα ή μένα από τους δε, αλλά οριζόντια σε διάφορους τομείς, προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια μεταξύ μόνη συνεργασία για να καταφέρουμε να προωθήσουμε συγκεκριμένες στρατηγικές. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα και θα ήθελα να διορθώσω κάτι το οποίο είπα. Ο κύριος Σεντσεβίτσιους, ο επίτροπος Σεντσεβίτσιους, δεν πρόφερα σωστά το όνομά του, είναι αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνο για τη στρατηγική για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Είναι στα πλαίσια δηλαδή της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες και όχι τόσο πολύ στο, στο, πλαίσιο της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο που θα αναλάβει ο επίτροπος αυτός δράση και προφανώς εγώ θα συνεργαστώ στενά μαζί του. Ας περάσουμε στην ε, τελευταίο, τελευταίο τρίτο γύρο ερωτήσεων, ξεκινώντας με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. κύριο Σάλκοβιτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, σε όλο τον κόσμο, ετησίως, έχουμε 450.000 φόνους και η αστυνομία διεθνώς έχει ένα σύστημα ε, δίωξης. Τώρα έχουμε τον καρκίνο. Δέκα εκατομμύρια θύματα του καρκίνου είναι παγκοσμίω. Έχουμε τα κονδύλια, έχουμε τις οργανώσεις και είναι καθήκον μας να ε, στήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα καταπολέμησης του καρκίνου. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα για έγκαιρη διάγνωση, για καλή πρόληψη, προφύλαξη, σύγχρονες θεραπείες προσπελάσιμες σε όλους. Οι πολίτες ε, το θέλουν αυτό πολύ, δεν θα μας συγχωρήσουν αν δεν το κάνουμε. Εγώ είμαι γιατρός και ογκολόγος. Το ένα τρίτο ε, από εμά που είμαστε εδώ παρόντες στην αίθουσα θα καταλήξουμε λόγω καρκίνου. Τώρα, να σας ευχαριστήσω για αυτό που είπατε. Δεν ξέρω αν πρέπει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κύριε Επίτροπε, είναι γνωστή πλέον η στρατηγική ε, από το αγρόκτημα στο πιάτο. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πολλέ προθέσει για τη μείωση των ζενοκτώνων, να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων και δημιουργούνται και νέε υποχρεώσει περιβαλλοντικέ για του γεωργού. Δηλαδή, περιορισμοί, απαγορεύσει, επιβαρύνσει. Ο τομέα τη γεωργία και ο γεωργιοτροφικό τομέα γενικά έχει όμω άλλε απαιτήσει οι οποίε επήγουν. Υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, υπάρχει ε, οργή ε, στου γεωργού. Ιδιαίτερα στην Ισπανία αυτή τη στιγμή, στην Εξτρεμαδούρα, ε, οι γεωργοί έχουν εξεθάψει το τσεκούρι του πολέμου. Ε, και αν δεν το αντιμετωπίσουμε αυτό, όλη αυτή η στρατηγική θα πάει στράφη. Ακούστε λοιπόν τους γεωργούς μας. Ακούστε τους γεωργούς όσο ακούτε και τους ιδεολόγους ε, των πόλεων. Ε, πώς ε, θα συμπεριλάβετε στη νέα στρατηγική επίσης πτυχές της εμπορικής πολιτικής για να μην έχουμε την εισαγωγή γεωργικών προϊόντων που περιλαμβάνουν όλα αυτά που θέλουμε εμείς να απαγορεύσουμε στην Ευρώπη. για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ είμαι αθλητίατρος. Ο προηγούμενος ήταν, ε, ο συνάδελφος ήταν ογκολόγος. Ε, και ο αθλητισμός παίζει ρόλο για τον καρκίνο. Όταν μιλάμε για τον καρκίνο πρέπει να πούμε ότι οι ανθυγιεινές συνήθειες είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου. Η ε, Ευρώπη επηρεάζεται από αυτό. Και το σχέδιο κατά του καρκίνου και το Farm to Fork μπορούν να μας βοηθήσουν να σώσουμε ζωές, να κάνουμε μια θετική διαφορά. Ο μέσος καταναλωτής αποφασίζει τι θα ψωνίσει πολύ γρήγορα. Οπότε το Nutri-Score είναι ένα πολύ καλό σύστημα όπου ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίσει με τρόπο απλό. Η επισήμανση Nutri-Score προτείνεται αυτή τη στιγμή από από κράτη-μέλη, δηλαδή 232 εκατομμύρια θέλουν πάνω από το μισό πληθυσμό της Ένωσης. Ε, γίνεται πολύ καλά αποδεκτό από τους καταναλωτές. Γι' αυτό ρωτώ, τι μπορούμε να περιμένουμε σχετικά όχι πότε, πότε εννοώ, πότε μπορούμε να περιμένουμε τη δημοσίευση της αξιολόγησης REFIT για τον κανονισμό σχετικά με τους ισχυρισμούς για υγιεινά τρόφιμα κλπ. Ευχαριστώ Επίτροπε για την ειλικρίνειά σας προς τα μέλη του Κοινοβουλίου και την Επιτροπή μας. Είπατε, εδώ είμαι, είπατε ε, ότι στα πλαίσια του Farm to Fork θα υπάρχουν και μέτρα για την καλή υγεία των ζώων. Επαναλαμβάνω για την Επιτροπή ότι στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου υπήρχαν δύο ε, παράγραφοι για την ε, καλή κατάσταση των ζώων που δεν ανταποκριθήκε η προηγούμενη Επιτροπή και για το ε, νόμο πλαίσιο. Αυτά έχουν ψηφιστεί με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, το Κοινοβούλιο δηλαδή θέλει τα δύο αυτά. Στην προηγούμενη θητεία κάναμε κάποιες καλές κινήσεις σχετικά με τη νομοθεσία για τα φάρμακα, αλλά και εκεί πρέπει να φροντίσουμε ότι θα διατηρηθεί η υλοποίηση. Ε, υπάρχει αντίσταση από κάποιες χώρες που και παλιά και τώρα ανθίστανται. Τώρα, Σουηδία, Νορβηγία. Ε, ε, βλέπουμε εδώ ένα προϊόν το οποίο απαγορεύεται στην Δυτική Ευρώπη και που εξετάζει ε, την μείωση του ρίσκου από κάπνισμα. Oui, merci, Madame la Je voudrais θέλω να επανέλθω στο θέμα της έλλειψη φαρμάκων στην Ευρώπη. 80% των ενεργών ουσιών παράγονται στην Ασία ε, λόγω του κορονοϊού αυξάνεται η ανάγκη. Ποιες είναι λοιπόν ε, ποια είναι τα μέτρα που παίρνετε για να αντιμετωπίσουμε την έλλειψη φαρμάκων στην Ευρώπη, το ίδιο και με το ιατροφαρμακευτικό υλικό και την, το προστατευτικό υλικό, τα, οι μάσκες που ε, τα μισά κατασκευάζονται στην Κίνα, όπου αυτή τη στιγμή έχουν έλλειψη. Υπάρχει το θέμα επίση τη συναρμόνιση του κανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο και των φαρμάκων και το πώ αυτά μεταφέρονται από ένα κράτο μέλο στο άλλο. Η πρόσβαση για όλους, στην υγεία για όλου του πολίτε πρέπει να εγγυάται με διαφάνεια σε ό,τι αφορά την διαθεσιμότητα των διαφόρων μορφών περίθαλψη. Πότε λοιπόν θα έχουμε ένα σύστημα ε, πληροφορική, ε, ειδικά για αυτόν τον σκοπό, για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά την τιμή των φαρμάκων, σε ό,τι αφορά το επίπεδο των. Ε, ε αποθεμάτων και άλλα χρήσιμε, άλλες χρήσιμες πληροφορίες ε, στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για την ΚΟΕ, ο Νίκου, Άλλας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν ε, μιλήσαμε για την υπερκατανάλωση και υπερπαραγωγή γαλακτοκομικών και κρέατος. Ε, υπάρχει ένα σχέδιο έκθεσης που δείχνει πολλές διαφορές. Η ό,τι αφορά λοιπόν την υπερκατανάλωση, μιλάμε για συστήματα βιώσιμης διατροφής. Η Κομισιόν έκανε στις 21 Ιανουαρίου μια παρουσίαση σχετικά με τη στρατηγική Farm to Fork και είπε ότι η μείωση των ζώων μπορεί να οδηγήσει σε ε, πρόβλημα βιοπικιλότητας. Τα δύο τρίτα όμως της αγροτικής γης αφιερώνονται στην κτηνοτροφία. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει να ναι, αποφύγουμε τις μονοκαλλιέργειες για την παραγωγή ζωοτροφών. Ε, πώς θα, θα γίνει ε, σωστή κτηνοτροφία με ε, σωστό αριθμό ε, ζώων εκτρεφωμένων και πώς μπορεί να αποφευθεί η υπερ ε, κατανάλωση και υπερπαραγωγή της εντατικής κρεοπαραγωγής. Λίζα ευχαριστώ. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την αξία επενεργασία που κάνετε. Πέρα από τις ανησυχίες που έχουμε και εμείς για τον Τρισκόρ, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πώς μπορούμε να είμαστε πραγματικά συνεπείς ε, όταν λέμε ότι θέλουμε να μειώσουμε τα φυτοφάρμακα, να αυξήσουμε τη βιωσιμότητα, ενώ έχουμε πάρα πολλά προϊόντα τα οποία μας έρχονται από τρίτες χώρες και τα οποία δεν συμμορφώνονται με τα δικά μας ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεύτερον, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, πρέπει να σας πω ότι ως ιατρός πρέπει να δούμε πώς η Ευρώπη μπορεί να καταπολεμήσει τον καρκίνο ενώ παράλληλα επιτρέπει την ε, διάθεση στο εμπόριο τροφίμων που περιέχουν πολύ επικίνδυνες καρκινογόνες ουσίες όπως για παράδειγμα τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Επίσης, πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη πρόσβαση από τους πολίτες εκείνους που δεν έχουν ε, τα απαραίτητα χρήματα στις απαραίτητες θεραπείες καθώς επίσης και στην απαραίτητη διάγνωση. Τελευταία από μία εγγεγραμμένου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αν, όπως λέτε, η Κομισιόν θέλει όντως να αλλάξει τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης τότε θα πρέπει να είναι πάνω από φιλόδοξη η στρατηγική ε, Farm to Fork. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τα, ε, ε, τις επιπτώσεις στο έδαφος, στον αέρα, στο υπέδαφος ε, κλπ. της εντατικής ε, γεωργίας και τις επιπτώσεις της μικροβιακής αντοχής όπως και τα δεινά των εκατομμυρίων ζώων που είναι αντικείμενα υπερεκμετάλλευσης παντού στον κόσμο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες μίλησαν ξεκάθαρα μέσα από τις πρωτοβουλίες των πολιτών. 1,6 εκατομμύρια ε, υπογραφές ε, ε, συγκεντρώθηκαν για να βελτιωθεί η καλή κατάσταση των ζώων. Η ΕΦΣΑ πρόσφατα έχει επίσης γνωμοδοτήσει για την καλή κατάσταση των ζώων και τονίζει ε, όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι γενικά η κατάσταση ε, είναι ε, καλή. Η Επιτροπή των Περιφερειών στη γνωμοδότησή της για την ΚΑΠ στηρίζει το αίτημα του να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται κλωβοί. Είναι μοναδική ευκαιρία λοιπόν να εξυγχρονίσουμε την απαρχιωμένη νομοθεσία για την κατάσταση των ζώων και ε, την εισαγωγή νέων συστημάτων για την εκτροφή ζώων. Ναι, εγώ θα πρέπει να φύγω και θα με αντικαταστήσει η πρώτη αντιπρόεδρος. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερος ε, και έχετε περίπου 10 λεπτά για να απαντήσετε στο τελευταίο γύρο. Thank you very much. Um, ευχαριστώ. Θα απαντήσω όχι με τη σειρά όμως. Πρώτα απ' όλα βεβαίως και ακούω τους γεωργούς. Πρέπει να ακούμε τους γεωργούς. Πρέπει να τους υποστηρίζουμε σε αυτή τη μεταβατική φάση. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να έχουν εναλλακτικέ που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους ε, και σε επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης, να βρεθούν εναλλακτικέ λύσεις βιώσιμης ε, ε, καλλιέργειας. Πρέπει να έχουν κίνητρα χρηματοδότησης για να μπορούν να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία μαζί μας. Και θέλω να είμαι σαφής. Στο πρόγραμμα ε, εκμετάλλευση από την εκμετάλλευση στο πιάτο θα έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για τον κίνδυνο χρήση ζανιοκτώνων. Με έχουν ρωτήσει πολλές φορές Έχω απαντήσει πολλές φορές Είναι σαφές λοιπόν. Τώρα, τα αποφάγια, όπως τα λέμε, γίνεται λόγο για δίαιτα και γη δίαιτα, γη διατροφή, ε, γίνεται λόγος. Θα πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το θέμα της πατάλης τροφίμων. Είμαστε, ε, ζούμε σε μια εποχή που δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε, σε μια γη διατροφή κάθε μέρα. Και παρόλα αυτά σπαταλούμε πολλά από αυτά τα τρόφιμα και θα πρέπει λοιπόν αυτό να το συμπεριλάβουμε στη στρατηγική μας, θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της βιώσιμης κατανάλωσης και να συζητήσουμε και το θέμα της υγιούς διατροφής, της υγιούς δίαιτας. Και αυτό έχει να κάνει και με την πρόληψη. Ο αξιοεξιολόγηση ρήφη τώρα, αυτή θα προκύψει ταυτόχρονα με το πρόγραμμα από την εκμετάλλευση στο πιάτο. Τώρα για την ευμερία των ζώων, βεβαίως πολύ σημαντικό ζήτημα, Γνωρίζω ότι αποτελεί προτεραιότητα το ζήτημα και ελπίζω ε, να ξαναδούμε την νομοθεσία αυτή ε, ως το τέλη του 2020, διότι πρέπει να την ξαναδούμε. Να δούμε λοιπόν τι θα αλλάξουμε και τι θα χρειαστεί τελικά να τροποποιηθεί. Ε, έλλειψη φαρμάκων. δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μία μόνο αιτία γι' αυτό. Όταν βλέπουμε το θέμα των φαρμάκων και τη πρόσβαση στα φάρμακα, πρέπει να δούμε ποιε είναι οι ελλείψει, ε, πρέπει να δούμε την τιμολόγηση, πρέπει να δούμε την, απο, την αποζημίωση. Ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Φαρμάκων εξετάζει αυτή τη στιγμή ε, τα ζητήματα αυτά. Αναμένουμε ε, την αξιολόγηση της σχετικής νομοθεσίας για τα ορφανά φάρμακα, να δούμε πώς μπορούμε ε, να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Σίγουρα θα μπορούσαμε να προβούμε σε κάποιες αλλαγές ε, και κάποιες αλλαγές τις οποίες μπορούν να προωθήσουν τα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε καλύτερες τιμές και μεγαλύτερα ποσοστά επιστροφής. Θα έχουμε μια στρατηγική για τα φάρμακα στο τέλος του 2020. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι και αυτό συνδέεται και με τον κορονοϊό και το προστατευτικό εξοπλισμό ήδη δεχτήκαμε αυτό που μας ζήτησαν τα κράτη-μέλη, δηλαδή κοινές, ε, κοινοί διαγωνισμοί ε, σε ό,τι αφορά την ε, απόκτηση τέτοιου εξοπλισμού. Το Nutri-Score τώρα, άκουσα προσεκτικά αυτό που ελέγχθη να μένουμε την έκθεση της Κομισιόν. Για την ώρα είναι θελοντικό αυτό το σύστημα. Θα πρέπει να πάμε προς μια εναρμόνιση βέβαια και θα επανέλθουμε με μια πρόταση επ' αυτού. Και για το Cage Age θα υποβληθεί το Σεπτέμβριο σχετική πρωτοβουλία. Από εκεί πέρα η Κομισιόν έχει 6 μήνες για να απαντήσει. Δεν μπορώ να σας πω ποια θα είναι η απάντηση. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι για μας είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και τέλος, Σας άκουσα πολύ προσεκτικά όταν αναφερθήκατε στον καρκίνο και τις 350.000 ε, ε, δολοφονίες ε, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είστε ογκολόγος βέβαια, έχετε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. έχω κι εγώ όμως εμπειρία καρκίνο, ξέρετε, και δεν χρησιμοποιώ λόγο που δημιουργεί φόβο και που στιγματίζει. Είναι ο καρκίνος μια ασθένεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Αυτό που είπατε λοιπόν για μένα είναι το, το πιο σημαντικό από αυτά που είπατε είναι ότι πρέπει να εργαστούμε πάνω στην πρόληψη. Να εργαστούμε για την πρόληψη με βάση όλα αυτά που υπόθηκαν σήμερα, διότι η πρόληψη δεν μπορεί να αφορά μόνο έναν τομέα της υγείας. Είναι οριζόντιο ζήτημα. Και όταν μιλάμε για το πρόγραμμα από την εκμετάλλευση στο πιάτο, εκεί η πρόληψη σίγουρα θα συνδέεται και με τη στρατηγική για τον καρκίνο. Μιλάμε για ασφαλή τρόφιμα και όταν μιλάμε για ε, φάρμακα και αυτό σχετίζεται με τη στρατηγική τα φάρμακα του 2020, διότι και αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση γύρω από τον καρκίνο. Συμφωνώ λοιπόν απολύτω μαζί σα, αλλά δεν ξέρω αν ήταν θέμα μετάφραση, αυτά συμβαίνουν καμιά φορά. Ε, δεν θέλουν να χρησιμοποιούνται όροι που δημιουργούν φόβο γύρω από τον καρκίνο, διότι ε, Μα πήρε πολύ χρόνο να μπορούμε να συζητούμε για αυτά τα πράγματα ανοιχτά. Πρέπει θετικά να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό για να φέρουμε την αλλαγή. Σα ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μα δώσατε, που μου δώσατε να είμαι εδώ σήμερα. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ την Επίτροπο θα τα βρείτε διμερό τα θέματα τα γλωσσικά και τον όρο που χρησιμοποιήθηκαν. Σα ευχαριστώ πολύ για τις σαφεί απαντήσεις σας. Νομίζω ότι απαντήσατε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα και αυτό είναι τιμητέο. Το Κοινοβούλιο αλλά και αυτή η Επιτροπή όλους διετέρως αναμένει την πρότασή σας ε, το Μάρτιο αλλά και τις υπόλοιπες προτάσεις. Μας ζητεί ε, η Επίτροπος να συνεχίσει να πιέζει η Επιτροπή μας και βεβαίω και θα το κάνουμε. 12 και μισή εδώ η ομάδα εργασία για την υγεία θα συνεχίσει τις εργασίες της ε, για τον καρκίνο, πολύ σημαντικό ζήτημα. Ξανά πίσω εδώ λοιπόν 2 και μισή για να ξεκινήσει η συνεδρίαση με την ψήφιση των αντιπροέδρων. Θα τα ξαναπούμε 2 και μισή λοιπόν εάν δεν είστε εδώ στην ομάδα εργασία για την υγεία.